Pas Καλώς ήρθατε στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία. Να σας εξηγήσω καταρχήν γιατί προεδρεύω εγώ. Ο βουλευτής ο οποίος προσωρινά ε, ασκεί την Προεδρία ε, πρέπει να είναι αυτός ο οποίος έχει εργαστεί περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει τις περισσότερες θητείες. Αυτό δεν σημαίνει, δεν σημαίνει βέβαια ότι είμαι ποιοτικότερο, αλλά είμαι πιο πολύ καιρό εδώ. Δεν με καταλαβαίνετε. Εντάξει, ακούτε τη διερμηνία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας θυμίσω ότι το αντικείμενο αυτής της συνεδρίασης είναι να δημιουργηθεί το Προεδρείο, το ειδικό Προεδρείο της, επιτροπής Το της Ειδικής Επιτροπής για την Θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο, στη συνέχεια έναν έως τέσσερις αντιπροέδρους, σύμφωνα με τα άθρα 197 και 204 του κανονισμού. Θα συσταθεί δηλαδή το Προεδρείο. Η σειρά με βάση αυτά που σας είπα είναι οι εξής. Πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο ή την πρόεδρο ελπίζω. Στη συνέχεια στους τέσσερις αντιπροέδρους και βεβαίως ε, για τις επόμενες εκλογές μετά την πρώτη, δηλαδή αφού εκλέξουμε τον πρόεδρο, θα προεδρεύει πλέον ο νέος πρόεδρος. είναι παρούσα εδώ και η γαλλική κρατική τηλεόραση France και θα μαγνητοσκοπήσει την ε, ε, συνάντησή μας είναι και πληρωτές τώρα που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία ε, να πω ότι οι πολιτικές ομάδες που έχουν προβεί σε αλλαγές θα πρέπει να ενημερώσουν, να με ενημερώσουν εμένα, δηλαδή τον προσωρινό πρόεδρο. Και αυτό πριν την ψηφοφορία. Εάν δηλαδή υπάρχει κάποια πολιτική ομάδα που αντικατέστησε μέλη της και δεν μας το έχει γνωστοποιήσει, πρέπει να το πράξει τώρα. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οι αναπληρωτές Συγγνώμη τώρα για τα ονόματα που θα τα πω εγώ. Κυρία Ντουμπράφκα, Σουίκα, αντικαθιστά την Άννα Μαρία Κοραζαμπίλ για το ΕΛΚ. Και ο κύριος Γιωζέπ Μαρία Νεκάμπρας ε, αντικαθιστά την Γιουντίτ Αργεντίνη για τους Πράσινους. Τώρα πρέπει να δω εάν υπάρχει απαρτία για την ψηφοφορία. Εν, το 1 τέταρτο δηλαδή των βουλευτών, 8 ε, δεν υπάρχει ζήτημα, δεν υπάρχει θέμα, η απαρτία υπάρχει. Λοιπόν, οι για την Προεδρία τώρα. Σας θυμίζω ότι οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν είτε από μια πολιτική ομάδα, είτε από το 1 εικοστό των μελών της Επιτροπής στην οποία περίπτωση δύο βουλευτές. Ε, οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων και οι υποψήφοι θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής. Επίσης, θα πρέπει όλοι οι υποψήφοι να έχουν κάνει τη δήλωση σχετικά με τα οικονομικά συμφέροντα. Έτσι ώστε να γίνουν όλα νομότυπα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να μου πείτε ποιοι είναι οι υποψήφοι. Ο κύριος Γερούν Λέναρτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εκ μέρου του ΕΛΚ. Την Ναταλή Γκρισμπέκ θέλω να προτείνω για πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Λενάρτς. Απευθύνομαι τώρα στην ε, κυρία Γκρίσμπεκ. Δέχεστε την υποψηφιότητα αυτήν. Ναι, βεβαίως ε, την δέχομαι. Δέχομαι να προεδρεύσω αυτής της Επιτροπής. Πολύ ωραία. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Όχι. Ο κανονισμός μας περίπτωση αυτή προβλέπει ότι η πρόεδρος θα εκλεγεί διαβοής. Ε, euh, Εγκαταλείπω λοιπόν αυτή τη θέση και δίνω το λόγο και την Προεδρία στη νέα Πρόεδρο την Αταλή Γκρισμπέκ. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου πριν περάσουμε στη συνέχεια της μέσα διάταξης να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Ε, είναι κάτι που με υποχρεώνει και μας υποχρεώνει γενικά ε, να σημειώσουμε πρόοδο για αυτό το σημαντικό ζήτημα, το λεπτό, απαιτητικό. Θα πρέπει λοιπόν να να υπάρξει ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και στα πλαίσια βέβαια των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Εάν δεν έχετε αντίρρηση θα περάσουμε τώρα ε, στην συνέχιση της ημερής διάταξης για να μπορέσουμε να ε, ολοκληρώσουμε τη σύσταση, του Προεδρείου αυτής της ειδική και προσωρινής επιτροπής. Θα εκλέξουμε τώρα λοιπόν διαδοχικά τους διάφορους αντιπρόεδρους. Ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες με αυτούς που ανέφερε ο Ζεράντο Πρέ προηγουμένως, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που προείδρευσε, ε, προείδρευσε για λόγους, λόγω του κανονισμού και για βιολογικούς λόγους, όπως περιπτώσει. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσω και εγώ τους ίδιους κανόνες για να εκλέξουμε τους τέσσερις αντιπροέδρους. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή ε, σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με προηγουμένως, εάν κάποια πολιτική ομάδα δεν μας έχει γνωστοποιήσει ε, κάποια αλλαγή να το πράξει τώρα. Ε, λοιπόν, η κυρία Ντουμπράσκα Σουίκα, λοιπόν, ε, αντικαθιστά την Αναμαρία Μαρία Κορατζαμπίλτ και ο κύριος Τζοζέπ Μαρία Κάβρας ε, αντικαθιστά ως αναπληρωματικό μέλος την κυρία Γιουντίτ Σατζεντίνη. Λοιπόν, απαρτία υπάρχει και τώρα θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι υποψήφιος για την πρώτη προεδρία. Ο κύριος Ντεπρέ έχει στήσει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. με μεγάλη χαρά εκ μέρους της ε, Άλντε προτείνω την ψηφιότητα του Γερούν Λέναρτς. Α, είναι η τρίτη αντιπροεδρία αυτή. Ναι, για την πρώτη αντιπροεδρία. Δίνω αυτή αμέσως το λόγο στην Άννα Γκόμες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και εξ ονόματο τη ομάδα μου θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα για την πρώτη αντιπροεδρία την κυρία Ελένα Βαλενσιάνο η οποία είναι αντιπρόεδρος στην ομάδα μας και έχει διτελέσει και Στην Αντιπρόεδρο στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βαλενσιάνο συμφωνεί με την υποψηφιότητα αυτή. Ναι, είμαι σύμφωνη και ευχαριστώ την ομάδα μου. Σας ευχαριστώ και να σα υπενθυμίσω τη συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία σε ό,τι αφορά την υπογραφή της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων και θα ήθελα να σας προτείνω αν δεν ζητείτε μυστική ψηφοφορία, να εκλέξουμε σε σύμφωνα με τον κανονισμό την πρώτη αντιπρόεδρο τη ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την κυρία Έλληνα Βαλανσιάνο. Και θα σα ζητήσω να έλθετε κι εσεί εδώ δίπλα μου ω πρώτη αντιπρόεδρο. Συγχαρητήρια εξ ονόματο όλη της επιτροπή μας. Euh, Γυναίκες ε, μόνο ως τώρα. αλλά πρέπει να υπάρχει και σωστή προσώπηση των ανδρών. Τώρα, να υποβάλουμε υποψηφιότητε για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Ζωζεφ Μαρία Τρακάμπρας. Σας στο ονόματο τη ομάδα μου θα ήθελα να προτείνω την κυρία Σαργεντίνη, Σαργεντίνη ως δεύτερη αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Σαργεντίνη. Έχει συμφωνήσει ήδη, έχει συνενέσει ήδη για την υποψηφιότητα αυτή στη θέση τη δεύτερη αντιπρόεδρου. Και η γραμματεία επίση έλεγξε την δήλωση οικονομικών συμφερόντων για την κυρία Σαργεντίνη. Προτείνω λοιπόν να την εκλέξουμε διαβοής και αυτήν. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυρία Σαρχεντίνη. Οι φίλοι της θα της ε, διαβιβάσουν λοιπόν το μήνυμα. Και τώρα έχουμε την υποψηφιότητα για την τρίτη αντιπροεδρία. Ο κύριος Ντανζόν έχετε λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, στη θέση της, του τρίτου πρόεδρου, θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Γερούν Λέναρτς, για να υπάρχει και λίγο ισότητα μεταξύ των φίλων. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντανζόν. Ο κύριος Γερούν Λέναρτ. δέχεται την υποψηφιότητα αυτή για τη θέση της τρίτης αντιπροεδρίας και όχι μόνο επειδή είναι άντρας. Με χαρά αποδέχομαι την υποψηφιότητα, μιας και είμαι ο υπεύθυνο για την ποσόστοση, να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μάλιστα. Με ενημερώνουν λοιπόν οι υπηρεσίε ότι και εσεί έχετε ε, υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και Διαβοής θα σας εκλέξουμε και εσάς, κυρία Γερούν Λενάτς. Έλατε κι εσείς ε, στο Προεδρείο. Σας ευχαριστώ και σε χαρακτηρία. Να περάσουμε λοιπόν στην τελευταία αντιπροεδρία. Τέταρτη θέση αντιπροέδρου. Η κυρία Στέβενς. Η Έλκα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να υποβάλω την υποψηφιότητα του κυρίου Τζέφρι Φανόρντον ε, ως ε, υποψήφιο για την τέταρτη αντιπροεδρία από το, την ομάδα των συντηρητικών και ε, μεταρρυθμιστών. Δέχεται ο κύριος Φανόρντον. Είστε μπροστά μου και δεν σας έβλεπα. Αποδέχεστε την υποψηφιότητα αυτή? Μάλιστα. Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα. Ελέγξαμε λοιπόν τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Αν όλοι συμφωνείτε, διαβοή εκλέχθηκε. Περάστε και εσείς εδώ στο Προεδρείο. Merci beaucoup. Euh, Σας ευχαριστώ όλους. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το δεύτερο σημείο της ημέρησιας διάταξης. Το τρίτο σημείο είναι οι ανακοινώσει της Προέδρου. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ σε ό,τι αφορά τη δημιουργία αυτής της προσωρινή Επιτροπής να πω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων για τους συνεισηγητέ τη ειδική επιτροπή μας που είναι η κυρία Μόνικα Ολμέγερ από το ΕΛΚ και η Έλγα Στίβενς. Ήθελα λοιπόν να ε, σας το γνωστοποιήσω. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις. Πολύ ωραία. Θα είναι δύσκολη αυτή η δουλειά, αλλά και συναρπαστική. Θα έχουμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε και μία έκθεση στα μέσα της θητείας μας. Θητεία η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο. Λοιπόν, για τις επόμενες εργασίες της Επιτροπής μας τώρα. Η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης της Επιτροπής θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή αργότερα, όσο γίνεται πιο γρήγορα βέβαια, όταν οι συντονιστές της κάθε ομάδας θα έχουν προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα συναντήσεων και βεβαίως το τι θα συζητηθεί εκεί. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Θα είναι ε, πολύ κοντά χρονικά οι συνεδριάσεις μεταξύ τους. Ελπίζω συντονιστές ε, να τα οργανώσουν καλά όλα αυτά. Θα έχουμε επισκέψεις, ακροάσεις, ε, και διάφορες εργασίες. Σας ευχαριστώ ε, για την επίοικια που δείχνεται σχετικά με την ημερομηνία αυτή την οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ε, η γραμματεία μου θύμισε άλλωστε ότι η επόμενη ημερομηνία εξαρτάται και από την, ε, ε τις υπηρεσίες διερμηνίας για να μπορέσουμε να εργαστούμε από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, δηλαδή με διερμηνία υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και από αυτού. Αυτά λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ. Όπως ε, ξέρετε άλλαξε και η ώρα της ψηφοφορίας, 11.30 έχει πάει. Ε, σας ευχαριστώ και καλή δουλειά μας σε όλους.